αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και σας καλωσορίζω όλους. Σας υπενθυμίζω ότι ο σκοπός της συνεδρίασης αυτής είναι η συγκρότηση σε σώμα και η ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρίου της Επιτροπής μας βάσει του άρθρου 213 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκλέγουμε πρώτα τον πρόεδρο και μετά θα εκλέξουμε τους αντιπροέδρους. Έχω αναλάβει εγώ την Προεδρία τώρα γιατί είμαι ο παλιότερος, όχι ο μεγαλύτερος ηλικία, ο παλιότερος. Δεν θα αλλάξουμε τώρα τις ημερομηνίες γέννησης. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι υπάρχουν κάποιοι αναπληρωτές. Τον κύριο, ο κύριος Ματζορίνο αντικαθιστά τον κύριο Λόπες, για παράδειγμα, στους σοσιαλιστές. Η κυρία Γκριγκόροβα θα αντικαταστήσει την κυρία Νόημαν από τους πράσινους. Ο κύριο Κάγκου θα αντικαταστήσει την κυρία Φωτίγκα στο ECR. Και κάποιος από την ID αντικαθιστά τον κύριο Μπακ, σωστά. Μπονφρίσκο, ο κύριος Μπονφρίσκο αντικαθιστά τον κύριο Μπακ και Άγγελα αντικαθιστά τον κύριο Φανόρντεν, σωστά. Και ο κύριος Ντεμάν αντικαθιστά τον κύριο Βλάσκο. Ωραία. Υπάρχει κάποιος άλλος αναπληρωτής, αν υπάρχει άλλη αντικατάσταση, πρέπει να το δηλώσετε πριν την ψηφοφορία. Σας ενημερώνω επίσης ότι υπάρχει ένα πακέτο καλωσορίσματος για όλους τους ευρωβουλευτές ε, στη θηρίδες σας. Και σας ενημερώνω επίσης ότι επειδή πρέπει να φύγω γρήγορα, θα με αντικαταστήσω ο κύριος Λόπες Ιστρικουάιτς για τη συνέχεια των διαδικασιών, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όσον με αφορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ζητώ από τη Γραμματεία να επαληθεύσει αν υπάρχει απαρτία. Να ξέρουμε πόσοι είμαστε πόσοι ψηφίζουμε. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω υπογράψει, αλλά φαντάζομαι ότι η γραμματεία μπορεί να μου φέρει τον κατάλογο εκεί για να υπογράψω και να φαίνεται ότι είμαι και εγώ παρόν εδώ. Υπενθυμίζω επίση ότι βάσει του άρθρου 218, για να έχουμε απαρτία πρέπει να έχουμε το 1 τέταρτο των μελών, δηλαδή 8 μέλη. Και με ενημερώνουν ότι έχουμε απαρτία. Ε? Μετρήσατε. Εντάξει, έχουμε παραπάνω. Καλώς. Υπενθυμίζω επίσης ότι ο υποψήφιος για την Προεδρία πρέπει να ορίζεται ή από το 5% των μελών της Επιτροπής ή από μια πολιτική ομάδα. Ότι θα υπάρχουν δύο ε, στην περίπτωση της ΕΝΤΕ. Και τώρα ζητώ υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου ή της Προέδρου. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μία υποψηφιότητα για την Προεδρία της ΕΝΤΕ. Ε, προτείνω την κυρία Ναταλή Λουαζό. Συμφωνείτε κυρία Λουαζό? Ναι, συμφωνώ. Ωραία, μια στιγμή, να σας είδα. Μια στιγμή. Η, η υποψήφια έχει τηρήσει τις υποχρεώσει τη. είναι δηλαδή τακτικό Για τη θέση προέδρου, έτσι, για την προεδρία τη ΣΕΝΤΕ και έχει υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων, οπω επιση και τον κώδικα θεατολογία. αλλε υποψηφιοτητε παρακαλώ. εσει Για τη θέση Προέδρου, έτσι, για την Προεδρία της ΣΕΝΤΕ. εν ονόματι του ID υποψήφιο προτείνω τον συνάδελφο Ζερόμ Ριβιέρ για τη θέση Πρόεδρου. The name is... Δεν έπιασα το όνομα. Ζερόμ Ριβιέρ. Ζερόμ Ριβιέρ. Ζερόμ Ριβιέρ. here. <laughs> Okay. Um, further nominations. Άλλες υποψηφιότητες παρακαλώ. Πρώτον, ο συνάδελφος συμφωνεί με την υποψηφιότητά του. Ναι, Πρόεδρε, δέχομαι με ιδιαίτερη χαρά την υποψηφιότητά μου. Έχετε κι εσείς ε, ολοκληρώσει τη διαδικασία ε, με την ε, δήλωση οικονομικών ε, συμφερόντων, όπως επίσης και με τον κώδικα διοντολογίας. Βεβαίως, όπως φαίνεται, εξάλλου διαδικτυακά στην σελίδα την διαδικτυακή. Ε, δεν την κοίταξα, ζητώ συγγνώμη, δεν κοίταξα την ιστοσελίδα στο ίντερνετ. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Ανώ. Πρόεδρε, έχουμε το προνόμιο, προνόμιο τέλος πάντων, να είμαστε μια από τις τελευταίες ε, επιτροπές που αποφασίζει σήμερα για το Προεδρείο της και διαπιστώσαμε ότι σε προηγούμενες ψηφοφορίες που έγιναν σε άλλες ε, επιτροπές δεν τηρήθηκε ο κανόνας don't. Κυρίως ε, μερικές φορές και σε βάρος των δικών μας υποψηφίων του ΕΛΚ. Οπότε για να αποφασίσουμε εδώ για τους υποψήφιους πρέπει να δούμε κατά πόσο οι υποψήφοι δέχονται να σεβαστούν τον κανόνα don't για τις υποψηφιότητες που θα ακολουθήσουν για τις αντιπροεδρίες στην Επιτροπή μας. Δεσμεύονται υποψήφοι υπέρ του συστήματος don't. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο να παρέμβει. Όχι από ό,τι βλέπω. Α, παρακαλώ κύριε Ριβιέρ. Πρόεδρε, ναι, επί τη ευκαιρία αυτή, ναι, θέλω να υπογραμμίσω ότι στο σύνολο των επιτροπών η ομάδα η δικιά μου, ε, ταυτότητα και δημοκρατία, αποκλείστηκε από το σύστημα αυτό DONT που σέβεται τις μειονότητες, οπότε πρέπει να πούμε ότι οι μειονότητες δεν γίνονται σεβαστές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξού και υποψηφιότητά μου. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση του μέλους του ΕΛΚ σχετικά με τις αντιπροεδρίες, εμείς δεν θα υποβάλουμε υποψηφιότητα για αντιπροέδρους. Πρόεδρος, πέρα από το σύστημα DONT που εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόστηκε, ο οποιοδήποτε υποψήφιο για την Προεδρία ή τις Αντιπροεδρίες πρέπει να έχει την πλειοψηφία της ε, υποπιτροπής μας. Οπότε ακόμα και αν υπάρχει το σύστημα τεχόντου, αν τα μέλη της Επιτροπής ή της Υποπιτροπής δεν τον ψηφίσουν και δεν έχει την πλειοψηφία, διαβοήση ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία, δεν προχωράει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Με μυστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Παρακαλώ, με το μικρόφωνο όμως. Είπατε ότι θέλετε να ρωτήσετε κάτι τους υποψηφίους, μα κανονικά δεν προβλέπετε. Επίσημα έχει υποβληθεί η υποψηφιότητά τους, έχουν καλύψει τις προϋποθέσεις. Δεν συνηθίζεται να γίνονται συζητήσεις με τους επιμέρους υποψηφίους. Λυπάμαι γι' αυτό. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε. Μυστική ψηφοφορία. Στο σύστημα θα εισάγουμε τα δύο ονόματα, σωστά. Λοιπόν, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ως εξή. Έχουμε δύο υποψηφίους, οπότε με τα δύο κουμπιά και το τρίτο της αποχής θα ψηφίσουμε. Ακούστε με λοιπόν προσεκτικά παρακαλώ. Η πρώτη υποψήφια ήταν η κυρία Λουαζό. Οπότε όσοι θέλουν να ψηφίσουν υπέρ της κυρίας Λουαζό θα πρέπει να πατήσουν το πράσινο κουμπί. Όσοι θέλουν να ψηφίσουν για τον κύριο Ριβιέρ θα πρέπει να πατήσουν το κόκκινο κουμπί. Και όσοι θέλουν αποχή θα πρέπει να πατήσουν το λευκό κουμπί. Λουαζό πράσινο λοιπόν. Ριβιέρ κόκκινο. Αποχή λευκό. Βάλτε την κάρτα σας στο μηχάνημα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Την έχετε? Εντάξει. Συνεπώς, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Και το μπλε κουμπάκι δείχνει, το φως δείχνει ότι είναι μυστική ψηφοφορία. Λείπουν τρεις ψήφοι εδώ. Τι συμβαίνει, δύο τώρα. Μα είμαστε στα μέσα τη ψηφοφορία. Ξέχασα την κάρτα μου στην άλλη αίθουσα που ήμουνα. Η γραμματεία έχει κάρτες για την ψηφοφορία. Να σας δώσει. Η γραμματεία έχει τέτοιες κάρτες να μοιράσει, οπότε θα σας δώσει. Όχι θα έπρεπε ο κάθε ευρωβουλευτή να φροντίσει να έχει την κάρτα μαζί του. Αλλά τώρα έχουμε 27 στους 27. Λίγη ψηφοφορία λοιπόν. Αποτέλεσμα. Α, λυπάμαι, για τεχνικούς λόγους κάτι δεν πήγε καλά. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Πράσινο για την κυρία Λουαζό. Πράσινο κουμπί για την κυρία Λουαζό, κόκκινο κουμπί για τον κύριο Ριβιέρ. Παρακαλώ και το λευκό είναι αποχή. Εντάξει, ξαναψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίστε. Πράσινο, λουαζό, κόκκινο, ριβιέρ, λευκό, αποχή. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Εγώ ψήφισα. Ποιος θέλει ακόμα να ψηφίσει λοιπόν. Δύο. Ένας τώρα λείπει. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει πέρα της ψηφοφορίας. 14 ψήφους πήρε η κυρία Λουαζό, 8 ο κύριος Ριβιέρ και 4 αποχές. Οπότε εσείς εκλεγήκατε κυρία Λουαζό, συγχαρητήρια. Και ελάτε εδώ παρακαλώ. Να καθίσετε στη θέση του Πρόεδρου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 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποδείξω ότι αξίζω την εμπιστοσύνη σας στην θέση εδώ της Προέδρου της Υποπιτροπής ΕΝΤΕ. Να ξέρετε ότι θα βασιστώ πολύ στην εμπειρία παλιότερων ευρωβουλευτών από εμένα θα βασιστώ δηλαδή πολύ σε ανθρώπους οι οποίοι όπω και εγώ έχουν δεσμευτεί και θέλουν να δουλέψουν για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλούς λόγους να έχουμε μια καλή συνεργασία μέσα σε αυτήν την υποεπιτροπή, αλλά και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σας λέω ότι εγώ δεσμεύομαι να ενισχύσω τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον τομέα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη ευκαιρία στη συζήτηση που θα κάνουμε με την κυρία Φόντερ Λάιεν... που είναι η υποψήφια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συνεχίζω στα γαλλικά, λέει η κυρία Λουαζό. Θα ακούσουμε επίσης και τον είπα το εκπρόσωπο και την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της. Και του χρόνου θα έχουμε και το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στην ατζέντα μας. Θα συζητήσουμε λοιπόν και για την πολιτική αυτή και ασφάλειας που ελπίζουμε να καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Δεν ε, πρέπει εδώ να ξεχάσω να σας πω τι λέει στο προήμιο η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για την πολιτική μας, μιλάει για μια κοινή πολιτική η οποία ενισχύει την ταυτότητα της Ευρώπης και την ανεξαρτησία της, προκειμένου να έχουμε ασφάλεια και πρόοδο στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο. Και μάλιστα σε μια στιγμή που όλοι το γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη ε, στιγμή. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια ειρήνης, αυτό είναι αλήθεια, από την άλλη μεριά ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσες πολλές και διαφορετικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και στα σχέσεις μεταξύ μας αλλά και με τρίτες χώρες και μέσα σε ένα γεωστρατηγικό πλαίσιο που όλοι το γνωρίζουμε είναι αρκετά ασταθές. Μέσα όμως σε ένα πλαίσιο επίση συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις χώρες μέλη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική και θα έλεγα και περισσότερο αποτελεσματική. Αυτά είναι τα καθήκοντά μας. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και ελπίζω να τις αντιμετωπίσουμε μαζί από κοινού. Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη και να περάσουμε στην εκλογή διαδοχικά των διάφορων αντιπρόεδρων. Δεν θα επαναλάβω την πληροφορία που σας έδωσα για τα αναπληρωματικά μέλη που αντικαθιστούν τακτικά, εκτός εάν μου πείτε ότι υπάρχει κάποια αλλαγή ανάμεσα στην ψηφοφορία που κάναμε για την Πρόεδρο και ε, τις αντιπροεδρίες. Αν υπάρξει αλλαγή να μου το πείτε απαρτία έχουμε. Οπότε, παρακαλώ, πείτε μου ποιες είναι οι υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ε, προτείνω τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη ως υποψήφιο για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Ο υποψήφιος αποδέχεται την υποψηφιότητα. Ναι, φυσικά την αποδέχομαι. Έχετε εκπληρώσει υποχρεώσεις όσον αφορά τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και το διντολογικά. Υπάρχουν άλλες ε, υποψηφιότητες για τη θέση πρώτου αντιπρόεδρου. Δεν βλέπω να υπάρχουν. Σας προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία διαβοής. Συγχαρητήρια και παρακαλώ να έρθετε εδώ στο βήμα. So now we will proceed with the... Uh, Περνάμε τώρα στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου. Ποιος θέλει να αναφέρει κάποια υποψηφιότητα, ο κ. Κυρία Πρόεδρε, για το ΕΛΚ προτείνω το συνάδελφο Κίντα Γκάλ. Yes. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, παρακαλώ. Ναι, ναι Πρόεδρε, δεν θέλω να, παρουσιάσω κάποια άλλη υποψηφιότητα. Απλώ ε, εκ μέρου των έξι παριστάμενων μελών του, των σοσιαλιστών ε, θα ήθελα να ζητήσω εδώ σε ό,τι αφορά την ε, θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου μυστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνά ε, με το καταστατικό μας ε, αφού έχετε έξι μέλη από την πλευρά της πολιτικής ομάδας που ζητούν μυστική ψηφοφορία αυτό θα γίνει. Μπορούμε λοιπόν να προβούμε σε μυστική ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καθώς υπάρχει μόνο μία υποψήφιος, εάν είστε, ψηφίσετε υπέρ, πατάτε το πράσινο κουμπί. Αν ψηφίσετε κατά, πατάτε το κόκκινο κουμπί. Και αν θέλετε να απόσχετε, να πέχετε μάλλον, θα πιέσετε το λευκό κουμπί. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. I close the vote. Πέραση τη ψηφοφορία. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Κυρία λοιπόν, ε, εκλέγεται, τη συγχαίρουμε και μπορείτε να έρθετε εδώ στο Προεδρείο. Συνεχίζουμε. Περνάμε στην εκλογή λοιπόν του τρίτου αντιπροέδρου. Υπάρχει κάποιος που θέλει να αναφέρει μια υποψηφιότητα. Ναι. Για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου προτείνω τον λέμε Ντεμιρέν. που μεγαλώσε στη Γερμανία και ήταν ο κορυφαίος υποψήφιος ε, της ε, D-Link εκ μέρους της ε, γερμανικής αντιπροσωπείας για την επιτροπή μας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. You accept your nomination. Αποδεχόμαστε λοιπόν, αποδέχεται μάλλον ο υποψήφιος αυτή την υποψηφιότητα, πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο υποψήφιο, α προχωρήσουμε λοιπόν σε εκλογή διαβόή. Σας συγχαίρουμε. Ελάτε και εσεί σας παρακαλώ στο Προεδρείο. Περνάμε στην εκλογή του τετάρτου Αντιπροέδρου. Ποιο θέλει να υποβάλει κάποια υποψηφιότητα, ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, ονόματι του ΕΛΚ, προτείνω τον κύριο Μάντελ, τον συναδελφό μου, για τη θέση αυτή. Μάντελ, do you accept the nomination? Αποδέχεστε την υποψηφιότητα, κύριε Μάντελ. Πολύ καλά. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε υποψηφιότητε. Προτείνω λοιπόν να επιβεβαιώσουμε την εκλογή του κύριου Μάντελ διαβοή. Σα συγχαίρω και ελάτε και εσεί στο Πρόεδρο... Ολοκληρώσαμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα της σημερινής διαταξής μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ανακοινώσεις της Προέδρου θα ήθελα να σας ε, αναφερθώ στο ζήτημα της ε, μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στο Προεδρείο σε ό,τι αφορά τη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Ε, με βάση λοιπόν το ε, άρθρο 214 του καταστατικού μπορεί ε, πέραν δηλαδή της υιοθέτηση της γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων να αναλυφθεί από την ομάδα των συντονιστών η αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων από κοινού με το Προεδρείο. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, θεωρούμε πως αυτή η απόφαση υιοθετείται, εγκρίνεται και από εκεί και μετά έχετε λάβει και ένα ημερολόγιο σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες συνεδριάσεις του 2019. Ε, Έχουμε λοιπόν τις εξής συνεδριάσεις. Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, ε, Σεπτέμβριο 25 και Σεπτέμβριο 26, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και Τρίτη 8 Οκτωβρίου, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, και Τρίτη 12 Νοεμβρίου και Δευτέρα Δεκεμβρίου, Δευτέρα και 3 Δεκεμβρίου, Τρίτη. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται και αυτές οι ημερομηνίες συνεδριάσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, το γλωσσικό καθεστώ σε ό,τι αφορά την υποεπιτροπή, ε, αυτό θα αποφασιστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση των συντονιστών της ε, ομάδας ΣΕΝΤΕ που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα. η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, θα λάβει χώρα στις 9 ε, Σεπτεμβρίου από τις 10 ε, στις 2.30. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για τη δουλειά τους και αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν τον λόγο, θα ήθελα να σα προτείνω να κλείσουμε εδώ τη συνεδρίασή μα και σα ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.